So, um, Καλησπέρα σας. Θα προεδρεύσω εγώ σε αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας διότι η πρόεδρος ε, θα έρθει κατά τις 5.30 είχε μια καθυστέρηση για την οποία δεν μπορούσε να κάνει κάτι στο ταξίδι της μια μισή ώρα λοιπόν καθυστέρηση και ζήτησε από του αντιπροέδρου να αναλάβουν κατά την απουσία τη. Πράγμα που θα κάνω. Και επειδή ξεκινάμε αργά τώρα το απόγευμα, θα ήθελα να προτείνω μια αλλαγή στην ημερήσια διάταξη, την ημερήσια διάταξη που έχετε παραλάβει, επειδή έχουμε προσκεκλημένου από το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα προσπαθήσουμε να μείνουμε στο χρονοδιάγραμμα αυτή τη παρουσίαση πιστή και το σημείο 5 να το δούμε πριν από το σημείο 4. 4 είναι η παρουσίαση της έκθεσης του κυρίου Χέτμαν. αν ε, μπορείτε να συμφωνήσετε λοιπόν στην ελλαγή αυτή, να εγκρίνουμε το σχέδιο μερίσης διάταξης για την ε, συνεδρίασή μας. Ερώτηση είναι αυτή. Κοιτώ τους συναδέλφους μου στα μάτια, δεν βλέπω να αντιδρά κανείς. Οπότε η μερίσια διάταξη με την αλλαγή αυτή εγκρίνεται. Δεύτερο σημείο, ε, έγκριση των πρακτικών της ε, συνεδρίασης 26 και 27 Μαρτίου 2018. Είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο και ως συνήθως, εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης, θεωρώ ότι εγκρίνονται. Δεν φαίνεται να υπάρχουν αντιρρήσει. Εγκρίνονται λοιπόν και περνάμε στο σημείο ακριβώ 5 τη ημερήσια διάταξη. Πολλοί είναι αυτοί που θα είδαν την έκθεση για το Κέντρο Γνώσεων και Επιστημών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κοινό ερευνητικό, την έκθεση που οργανώθηκε στο Στρασβούργο στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Στην έκθεση υπήρχαν 10 στάντ, εκ των οποίων ένα ε, ήταν αφιερωμένο στην ε, περιφερειακή πολιτική. Πολλά άλλα όμω έχουν επίση να κάνουν με τη δουλειά τη Επιτροπή μα. Με χαρά λοιπόν υποδέχομαι στη συνεδρίασή μα την κυρία Εμμανουέλα Μπελάν, που είναι διευθύντρια Ινστιτούτο για τι Διεθνεί σχέσει και την μονάδα Outreach του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου. Θα μα μιλήσει για το ρόλο του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου στην παροχή ε, βοήθεια και στήριξη προ τι εθνικέ, τοπικέ και περιφερειακές αρχές ε, για να μπορέσουν να κάνουν τι σωστέ επιλογέ στην περιφερειακή πολιτική και επίση για την πρωτοβουλία η επιστήμη συναντά τα κοινοβούλια του Ερευνητικού Κέντρου. Η κυρία Μπέλαν λοιπόν θα έχει πρώτη το λόγο για μια παρουσίαση 15 ε, λεπτών και μετά θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους για ερωταπαντήσεις. Έχουμε περίπου στις 5 για το σημείο αυτό. Κυρία Μπέλαν, έχετε το λόγο. Α, εκεί είστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και που προσκαλέσατε το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο να παρουσιάσει το έργο της σε αυτή την ε, διακεκριμένη ε, ομάδα βουλευτών. Ευχαριστίες και προς τους διερμηνείς Να δω αν δουλεύει αυτό. Ωραία λοιπόν. Είμαι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο αυτής. Είμαστε μια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για να πάω πιο γρήγορα Βιάστηκα λίγο. Μια πολύ σύντομη ε, ιδέα για την ε, αποστολή του κοινωνικού Κέντρου. Είναι το κέντρο επιστημών και γνώσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε γενική διεύθυνση, είμαστε μια υπηρεσία. Ε, ιδρυθήκαμε πριν από 60 χρόνια. Γιορτάσαμε την επέτειο των 60 ετών πέρσι για την ενασχόλησή μας με τις επιστήμες, ως επιστημονικό κέντρο δηλαδή από τα πυρηνικά ως ένα πολύ ευρύ θέμα θεμάτων που καλύπτουμε. Επενδύουμε στην διαχείριση γνώσεων και προγνωμοσύνης και αποστολή μας είναι να προσφέρουμε στήριξη στους ε, πολιτικούς ηθήνοντες, κυρίως όσους λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεργαζόμαστε με πάνω από 20 υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίσης, αυτό είναι σημαντικό στο συγκεκριμένο πλαίσιο, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε και να υποστηρίξουμε την, ε, ε, τον σχεδιασμό πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Προσφέρουμε επιστημονική στήριξη. Μας ε, δεσμεύει βεβαίως η επιστημονική μέθοδος, γιατί δεν έχουμε πολιτικές προτεραιότητες και είμαστε ανεξάρτητοι και επίσης εργάζομαι, εργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα ε, της ε, πολιτικής. 30% δεν είναι η σωστή παρουσίαση αυτή. 30% ε, της δουλειάς μας αφορά την προπαρασκευή της πολιτικής και το 40% την υλοποίηση αυτής. Εκεί εργαζόμαστε περισσότερο σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, διότι περισσότερη από την εφαρμογή της υλοποίησης της ευρωπαϊκής πολιτικής γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Ανέφερα τη γνώση, τη διαχείριση της γνώσης, knowledge management, Και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι σήμερα είναι απαραίτητο να παράγουμε γνώση και επιστήμη, αλλά υπάρχει τόσο πολύ στον κόσμο που το πιο σημαντικό είναι να δούμε από το τεράστιο αυτό όγκο γνώσης που υπάρχει γενικώ τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει τα κέντρα γνώσης που είναι ε, hub, κόμβι στο διαδίκτυο για να μπορέσουν ε, να τα αξιοποιήσουν οι χρήστε. Πολιτικοί θύνοντε από άλλε γενικέ διευθύνσει και επιστήμονε εκτό Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ε, εντολή να ε, πιστοποιήσουν τι γνώσει που υπάρχουν επί ενό συγκεκριμένου θέματο αλλά να είναι και εύληπτες οι γνώσεις που προσφέρουμε και αξιοποιήσιμες από τους πολιτικούς ευθύνοντες. Θα ήθελα εδώ περισσότερο να αναφέρω το κέντρο γνώσης για τις περιφερειακές πολιτικές, τις εδαφικές πολιτικές. Βλέπετε εδώ τα κέντρα που έχουν δημιουργηθεί. Ε, το πρώτο είναι από το 2015. Το 2016 έχουμε το κέντρο γνώσης για τις εδαφικές πολιτικές. Θα επανέλθω σε αυτά αργότερα. Μερικά παραδείγματα δίνουμε στήριξη στα κράτη-μέλη και τις ε, περιφέρειες. Γιατί είναι αυτό ενδιαφέρον για σας, γιατί είναι καλό να συνεργαστούμε. Γιατί για μας είναι ενδιαφέρον και σημαντικό να συνεργαζόμαστε με πολιτικούς ευθύνοντες, με τις περιφέρειες και τις πόλεις, τα αστικά κέντρα, διότι κατά αυτόν τον τρόπο παραμένουμε συνδεδεμένοι με την πραγματικότητα και με το πώς υλοποιούνται οι ευρωπαϊκές πολιτικές στην πράξη και έχουμε και αντίδραση για το πώς οι πολιτικές ε, εφαρμόζονται στην πράξη. Για τις περιφέρειες αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε είναι ένα τεράστιο φάσμα δεδομένων, πληροφοριών, επιστημονικών γνώσεων και δυνατοτήτων για την κατάρτιση μοντέλων, ε, δυνατοτήτων διαδικτύωσης, ανταλλαγής ε, βέλτιστων πρακτικών. Ο στόχος είναι πάντοτε να δίνουμε στους πολιτικούς ηθήνοντες επιτόπου γνώσεις και πληροφορίες ώστε να μπορούν ε, στο τέλος να προσφέρουν καλύτερη ε, πολιτική δράση για τους πολίτες. Λόγου χάρη. Ένα άλλο παράδειγμα. Η πλατφόρμα για τα ε, δεδομένα αστικών κέντρων. Αυτό είναι μέρος των εργαλείων που προσφέρουν τα κέντρα γνώσης. Τα κέντρα γνώσης που ανέφερα προηγουμένως. Κέντρο γνώσης για τις περιφερειακές πολιτικές συγκεκριμένα. Αυτό το κέντρο γνώσης προσφέρει υποστήριξη και βοήθεια σε περιφέρειες και πόλεις ώστε να υλοποιήσουν να ορίσουν, να υλοποιήσουν και να αναθεωρήσουν τις στρατηγικές τους για την ευθύ ε, εξειδίκευση. Θα γνωρίζετε προφανώς την ευθύ εξειδίκευση. Είναι μια προσέγγιση που βασίζεται στο επίπεδο το εδαφικό ε, για να καθοριστούν στρατηγικές που μπορούν να αξιοποιήσουν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες μιας συγκεκριμένη περιοχής, ενός συγκεκριμένου χώρου, γεωγραφικού χώρου και να αξιοποιήσουν τη διαδικασία της επιχειρηματικότητας όπου συμμετέχουν όλοι ε, και κυρίως πολιτικοί θύνοντες, επιστημο... Ε, καθηγητές πανεπιστημίων, ενδιαφερόμενοι για να καθορίσουν τι ανάγκε και τα ωφέλη που θέλει να αποκομίσει μια τοπική κοινότητα για να στοχεύσουμε καλύτερα τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Το κέντρο γνώση προσφέρει μια σειρά από εργαλεία και μηχανισμού συμβουλευτικής. Να ένα από αυτούς είναι χρήσιμος για τις αστικές περιοχές. Αυτό που βλέπετε είναι ακριβώς αυτό που εμφανίζεται και στον ιστότοπο ένα ωραίο γράφημα, μια γραφική αναπαράσταση των δεδομένων για τις πόλεις. Και βλέπετε δεδομένα για την οικονομία, την τοπική ανάπτυξη, τις μεταφορές, το περιβάλλον και πολλά άλλα. Και μπορείτε να τα ε, συμβουλευτείτε ανα πάσα στιγμή. Αυτό δίνει πληροφορίες στους πολιτικούς ηθήνοντες και τους πολίτες στην ανάπτυξη μελλοντικής πολιτικής. Αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα. Ο Άτλαντας. Ο Άτλαντας ATM,5. Ε, πέμπτη έκδοση, ανάλυση 800 αστικών περιοχών ε, που επιτρέπει να καταλάβουμε καλύτερα τους ε, τις πηγές παραγωγής σε κάθε γεωγραφική ομάδα. Μπορεί να βοηθήσει τους τοπικούς πολιτικούς ηθήνοντε να καταλάβουν καλύτερα ποιε είναι οι πηγές ρήπανση σε μια πόλη λόγου χάρη στην ίδια την πόλη ή από τις γειτονικές της περιοχές. Φταίνε οι μεταφορές, φταίει η θέρμανση, ε, η γεωργία. Αυτό είναι ένα εργαλείο για να στοχεύσουν καλύτερα τις πολιτικές τους και να μπορέσουν να ε, ε, αναλάβουν δράση και να επιλύσουν το πρόβλημα. Η ενεργειακή απόδοση, ένα άλλο εργαλείο που περιλαμβάνεται ως μέρος της πλατφόρμας αυτής για την ευφυή εξειδίκευση. Έχει να κάνει με την ενέργεια. Η ενέργεια, η θέρμανση δηλαδή, ο κλιματισμός, Αυτά ε, αφορούν το ίμιση της ε, ρήπανσης, είναι το ίμιση των πηγών ρήπανσης της πόλης συνήθως. Η πλατφόρμα μπορεί να βοηθήσει τους τοπικούς ε, ευθύνοντες να εντοπίσουν λύσεις ενεργειακής απόδοσης και να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να κινηθούν προς μια καθαρότερη ανάμειξη ενεργειακής πολιτικής για τις πόλεις. Είναι ένα άλλο παράδειγμα για το τι προσφέρουμε. Η ανθεκτικότητα, η αντοχή είναι ένα άλλο θέμα επίσης μεγάλη σημασία. Αυτό είναι ένα μοντέλο, ένα γράφημα που έχουν αναπτύξει οι επιστήμονές μας και εν μέρη βασίζεται σε γεωγραφικά δεδομένα αλλά έχουμε συμπεριλάβει και μαθηματικά στοιχεία συνεργαζόμενοι με τοπικές αρχές, λόγω χάρη με την πόλη του Μιλάνου. Οι επιστήμονε μας μπορούν να βοηθήσουν τους πολιτικούς ευθύνοντε σε τοπικό επίπεδο να ε, αξιολογήσουν την αντοχή των τοπικών υποδομών, των τοπικών υπηρεσιών, τι ενδεχόμενε ε, διακοπέ και αναταράξει για να βελτιώσουν τη μελλοντική του ε, αντοχή. Να ένα ακόμη εργαλείο, πολύ πρόσφατο, το οποίο παρουσιάστηκε και σε άλλη επιτροπή εδώ στο Κοινοβούλιο, το εργαλείο ελέγχου για την πολιτιστική ανάπτυξη των πόλεων. Είναι ένα διαδραστικό εργαλείο που αφορά περίπου 180 πόλεις νομίζω και δίνει ε, ενδείξεις και στοιχεία για την οικονομία και το ρόλο που μπορεί να έχει στην οικονομία η πολιτιστική διάσταση, η πολιτιστική παραγωγή των πόλων, ε, μουσεία, θέατρα, ε, είναι πάλι ένα εργαλείο που μπορούν να αξιοποιήσουν οι πολίτες, η, τοπική διοίκηση, οι πολιτικοί ευθύνοντες τοπικά, για να συγκρίνουν το πώς λειτουργεί η Ρώμη, ας πούμε, με άλλες παρόμοιες πόλεις, παρομοίων διαστάσεων. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι Είδαμε μετά την οικονομική κρίση ότι οι πόλεις που είχαν πολύ πλούσια πολιτιστική ε, οικονομία και οικονομία βασισμένη στη δημιουργικότητα άντεξαν καλύτερα στους κραδασμούς της κρίσης. Άρα μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευση και να βοηθήσει. Αυτό είναι ένα πυροελάχιστο τμήμα του συνόλου των ε, εργαλείων και στοιχείων συμβουλευτικής και πληροφοριών και μηχανισμών που μπορούμε να προσφέρουμε. Οπότε γι' αυτό και στο τραπέζι στην είσοδο έχουμε αφήσει τα διάφορα εγχειρίδια που παράγει το κέντρο. Το πρώτο έχει ένα κατάλογο ε, διεξοδικό όλων των εργαλείων που παρέχει το κοινό κέντρο. Το άλλο αφορά συγκεκριμένα την περιφερειακή διάσταση. Εάν σας ενδιαφέρει παρακαλώ να έρθετε σε επαφή μαζί μας και με χαρά να ε, προχωρήσουμε σε συνεργασία. Αυτό που θα θέλω να παρουσιάσω τώρα είναι η πιο πρόσφατη, η τωρινή μας πρωτοβουλία, που είναι η επιστήμη συναντά τα κοινοβούλια και η επιστήμη συναντά τι Περιφέρειες. Αυτό είναι ένα πολιτικό πρόγραμμα που το κοινοβούλιο ε, ευγενικά προσφέρθηκε να εγκρίνει. Ένα εκατομμύριο. Βασίζεται σε πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε το 2015 η οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο εδώ στις Βρυξέλλες και μετά προχώρησε και εκτός. Τη λανσάραμε και την εφαρμόσαμε σε συνεργασία με τοπικά και περιφερειακά κοινοβούλια. Το πιλωτικό πρόγραμμα μόλις εγκρίθηκε και μόλις πήραμε και την σχετική δημοσιονομική απόφαση και θα έχουμε τρεις βασικές δράσεις. Η πρώτη είναι 600 χιλιάδες ευρώ στοχευμένα για την ε, ε, πρωτοβουλία αυτή σε τοπικά συμβούλια, πόλεις και κοινοβούλια για το επιστήμη συναντά τα κοινοβούλια και επιστήμη συναντά της πόλης θέλουμε να βρούμε χώρους ε, και ομάδες όπου οι πολιτικοί θύνοντες και επιστήμονες μπορούν να συναντηθούν και να έχουν διάλογο το ιστορικό εδώ είναι η πηγή έμπνευση είναι διπλή οι ψευδείς ειδήσει, ο πολιτικός ε, λόγος που αλλοιώνεται από δεδομένα ψευδή, από απόψεις που δεν έχουν εξακριβωθεί, που ε, από το γεγονός ότι δεν υπάρχει συμφωνία σε ένα πραγματικό γεγονός για να καταρτιστεί μετά η πολιτική. Επίσης πώς οι επιστήμονες να έρθουν σε επαφή με πολιτικούς. Αυτά είναι θέματα στα οποία είμαστε ευαίσθητοι και εκεί θέλαμε να προβλέψουμε μια ευκαιρία, μια δυνατότητα να συναντηθούν οι πολιτικοί με τους επιστήμονες και ίσως μακροπρόθεσμα να διοργανωθεί ένα φόρουμ διαρκείας για να μπορεί αυτή η συζήτηση, αυτός ο διάλογος να έχει εξέλιξη. Έχουμε εντοπίσει θέματα για να συζητηθούν σε αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά το πιο σημαντικό για μας είναι το ζήτημα που επιλέγει να είναι ε, ενδιαφέρον και σημαντικό για τους πολιτικούς συνόντε σε τοπικό επίπεδο. Ας πούμε, το μέλλον της ε, περιοχής που παράγει κρασί μέχρι το περιβάλλον, την οικονομία, αυτό που πραγματικά ενδιαφέρει τους τοπικούς ηθήνοντες. Να πάω λίγο πίσω. επιλέξιμοι φορείς είναι τα εθνικά κοινοβούλια, τοπικά, περιφερειακά, είτε είναι κρατήδια της Γερμανίας, Λέντερ ή οτιδήποτε άλλη διοργάνωση έχει το κάθε κράτο, είτε σε επίπεδο πόλη κάποιο συμβούλιο. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να χρηματοδοτήσουμε μια τέτοια εκδήλωση και σχετικές μελέτες για το ζήτημα που θα απασχολήσει την εκδήλωση. Μελέτες οι οποίες μπορεί να εκπονηθούν πριν την εκδήλωση για να δώσουν τροφή για τη συζήτηση ή να προκύψουν μετά την ε, εκδήλωση για τη μελλοντική πολιτική δράση. Οι περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα και τις ενθαρρύνουμε θερμά να ε, οργανωθούν σε ομάδες ε, δύο πόλεων ή περισσότερων για να συζητήσουν ένα θέμα που ενδιαφέρει πολλούς ταυτόχρονα. Για μια πόλη που μπορεί να έχει μια λύση να προτείνει μια περιφέρεια, είναι επίσης ενδιαφέρον για τους υπόλοιπους να την ακούσουν και αυτές οι εκδηλώσεις, τέλος πάντων προχωράνε μόνο στους εγκεφάνειες, οι περιφέρειες μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να ε, διασυνδεθούν. Τελευταίο και πολύ γρήγορα, υποδομές έρευνας, απλώς ε, προς ενημέρωσή σας. Το κοινό κέντρο ερευνάς έχει ε, καταστάσεις και έδρα στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιταλία, τις κατοχώρες και την Ισπανία, σε πέντε χώρες. Στα επιτελεία μας αυτά έχουμε 69 ερευνητικά ε, εργαστήρια υποδομές, που είναι από το πιο απειροελάχιστο μέχρι το γιγαντιαίο πυρηνικό κέντρο έρευνας. Μια άλλη πρωτοβουλία είναι το να ανοίξουν οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις αυτές σε επιστήμονες ή ακόμη και επιχειρήσεις των κρατών μελών και ε, συνδεόμενων χωρών. Να προχωρήσουμε εδώ λίγο, επόμενη διαφάνεια. η πρόσβαση αυτή μπορεί να οργανωθεί ανάλογα με το ενδιαφέρον των ε, διαφόρων συμμετεχόντων. Δηλαδή κάποιος να έρθει να μας ζητήσει ε, από εμά το ερευνητικό κέντρο με χαμηλότερο κόστος να έχει πρόσβαση, αλλά είμαστε ανοιχτοί και στο χώρο των επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσει κάποια επιχείρηση να οργανώσει δοκιμέ και πειραματισμού για να ε, σχεδιαστούν νέα προϊόντα και να ε, ευνοηθεί και η οικονομική παραγωγή. Με αυτά βλέπετε τον, ιστότοπο, τον κατάλογο των κέντρων που μπορείτε να τα δείτε ε, και κλείνοντας να σας ευχαριστήσω και πάλι που με προσκαλέσατε και να σας παρακαλέσω με κάθε τρόπο Εάν κάτι από αυτά που είπα ή κάτι που σας φαίνεται ενδιαφέρον από όσα διαβάσατε στα φυλάδια μας, στα εγχειρίδια, ε, ή σε εσά ή στους ε, ψηφοφόρους σας, ε, τους πολίτες, να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Γιατί η πρωτοβουλία αυτή, το πολιτικό πρόγραμμα, είναι κάτι που ενέκρινε το Κοινοβούλιο και ανυπομονούμε να την εφαρμόσουμε. Και να έχει και συνέχεια, να έχουμε εκδηλώσει ή δυνατόν σε όλα τα κράτη-μέλη. Με κάθε λοιπόν ε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω με κάθε σεβασμό να την ε, διαβάσετε και να σας πω ότι έχουμε υποβολή για την προσφορά ενδιαφέροντος online. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπέλα. Οι συνάδελφοι μήπως έχουν ερωτήσει να υποβάλλουν στην καλεσμένη μας. Θέλει κάποιος συνάδελφος μήπως το λόγο. Ο κύριος Μπόγκοβιτς πολύ σημαντικό, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρώπη. Με ενδιαφέρουν τρία πράγματα. Πρώτον, ε, μπορείτε να μας πείτε κατά πόσο υπάρχει κάτι ανάλογο σε κάποιο άλλο σημείο του κόσμου στην Ευρώπη. Και έπειτα πόσο σημαντικό είναι αυτό όσον αφορά το έργο της ε, Κομισιόν ε, κατά την εκπόνηση του νέου πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου. Επίσης, υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ χωρών μελών, δηλαδή αξιοποιούν οι χώρες μέλη την ανταλλαγή δοκισμένων πρακτικών και τη χάραξη στρατηγικών περιφερειακών και κατά πόσο σε, οι μικρές κοινότητες έχουν ε, πρόσβαση ε, σε σχέση με την ε, συζήτηση που γίνεται για την περιφερειακή ανάπτυξη στα σχολεία κλπ. Γίνεται μια σχετική έρευνα. Σας ευχαριστώ. Και εγώ έχω μια ερώτηση για την ανταλλαγή πληροφοριών όχι μόνο μεταξύ των δήμων ή των πόλεων, αλλά και μεταξύ οργανώσεων που δραστηριοποιούνται εκεί, στους δήμους ή τα αστικά κέντρα. Δεύτερη ερώτηση. Γιατί έχετε γραφεία μόνο σε λίγες χώρες, μόνο σε πέντε χώρες και όχι σε όλες. Ειδικός λόγος γι' αυτό. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς παρακαλώ. Δεν βλέπω κανένα, οπότε να θέσω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Με ποια κριτήρια εφαρμόζετε τη στρατηγική σας και με ποια κριτήρια διαλέγετε τα θέματα, το ότι εγκύπτετε σε συγκεκριμένα θέματα στο κέντρο σας και αν ναι, ποια είναι αυτά τα κριτήρια. Ελά. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής για τις απορίες τους. Θα κάνω ό,τι μπορώ, θα βάλω τα δυνατά μου για να απαντήσω. Ως προς την πρώτη ερώτηση της δημόσια διοίκηση, στη διοίκηση Ευρωπαϊκή Επιτροπής και είμαστε ερευνητικό κέντρο, κάτι που μας προσδίδει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πάντως, με πανεπιστήμια, με περιφέρειες, με κράτη-μέλη, με το Υπουργείο Έρευνας ενός κράτους μέλους για παράδειγμα. Τα κριτήρια είναι συνήθως η επιστημονική αριστεία και η κοινότητα του αντικειμένου προς έρευνα. Περίπου 100 νέες συμφωνίες ε, επιστημονικής συνεργασίας το χρόνο συνάπτουμε και μάλιστα τα πορίσματα των ερευνών αυτών τα δημοσιεύουμε από κοινού με ένα ευρύ οργανώσεων. Οπότε δεν έχει νόες και κέντρα. Γιατί σε ό,τι αφορά την ευφύ e, ειδίκευση, για παράδειγμα, στο τομέα της ευφύης e, ε, ειδίκευσης ε, έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία στην Ευρώπη. Είναι υποχρεωτικό αυτό το θέμα στην Ευρώπη. Και επίση σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τις περιφέρειες, η πλατφόρμα για την ΕΦΑ, στοιχεία, τα δεδομένα τη πλατφόρμας αυτή. Και αυτή τη στιγμή τα μισά κράτη-μέλη και περίπου 180 περιφέρειες έχουν εγγραφεί και έχουν πρόσβαση και στενή ε, ενεργό συνεργασία με εμά για θέματα ευφυού ειδίκευση. Ταυτόχρονα όμω έχει εκδηλωθεί σοηρό ενδιαφέρον η Αμερική. Και μάλιστα φέτο το, φθινόπωρο θα έχουμε στη Σεβίλη μία ε, διάσκεψη με ευρύτερη συμμετοχή και έτσι θα προσπαθήσουμε να προβάλλουμε και να εξαγάγουμε κατά κάποιο τρόπο το ευρωπαϊκό μοντέλο. Μικρότερε πόλει, οι κομοπόλει, πώ ε, έχουν δεχτεί τα σχέδιά μα και τι μελέτε μα, εξαρτάται από το θέμα κάθε φορά. Θέματα όπω η εφήση, η δίκευση δημιουργούν ε, συνεργασία με πολλούς ε, αντισυμβαλόμενους, με πολλές περιφέρειες, δήμου. Αυτή η συνεργασία θα ενταθεί στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή των πληροφοριών. Σας είπα ότι έχουμε πολλές συμφωνίες με εταίρους. Τώρα, γιατί έχουμε παραρτήματα μόνο σε πέντε χώρες. Ίσως δεν έδωσα σωστές εξηγήσεις. Δεν είναι τα γραφεία αυτά ξεχωριστά. Είναι τμήματα των το, το γραφείων, γιατί έχουμε γραφεία στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο και στην Ίσπρα που είναι Το μεγαλύτερο μας ερευνητικό κέντρο είναι το τρίτο μεγαλύτερο κέντρο της Επιτροπής ό,τι φορά το προσωπικό που απασχολείται εκεί. Οπότε ανήκει γέννη στην έδρα, στο αρχηγείο μας. Ε, βέβαια, τέτοια παραρτήματα το κέντρο μας έχουμε σε πέντε χώρες και καταρχήν το Κοινό Κέντρο Ερευνών ασχολούνται με πυρηνικές ε, μελέτες. Οπότε οι περισσότερες ε, καταστάσεις ήταν πυρηνικές, βέβαια παραπλησμένες ως προς το πυρηνικό του έργο, αλλά η αρχή έγινε από τα πυρηνικά θέματα, από, την έρευνα για τα πυρηνικά θέματα και που μελετούμε. Επαναλαμβάνω, το Κοινό Κέντρο Ερευνών είναι ανεξάρτητο ως προς την επιλογή των επιστημονικών μεθόδων του. Αυτό ισχύει αλλά τικών που ασχολούνται με συγκεκριμένου τομεί εν ώψη της χάραξη πολιτικών στους συγκεκριμένους τομείς ή προκειμένου να εφαρμοστεί η νομοθεσία στους πρόγραμμά μας σε αιτήσια βάση. Ελπίζω να απάντησα στις απορίες σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπέλαν. Ε, ε, διαμορφώνεται, προσπαθείτε να διαμορφώσετε την κοινή γνώμη, προβάλλετε το έργο σας προς τα έξω. Ε, υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης προβολής ναι, ε, η απάντηση είναι ναι, προσπαθούμε να το κάνουμε. Ε, βεβαίως, έχουμε μια σχετική στρατηγική επικοινωνίας και απευθυνόμαστε σε διάφορα τμήματα των ψηφοφόρων, με επιστήμονες, ε, με τους ευθύνοντες της πολιτικής και βεβαίως το κοινό. Για παράδειγμα, έχουμε Επίσης στην Ιταλία, στην Ίσπα, ένα κέντρο επισκεπτών όπου οι πολίτες μπορούν να το επισκεφθούν, να πειραματιστούν και να δουν ε, το έργο μας ε, σε πραγματικό χρόνο. Καλύφθηκε η ερώτησή σας. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπελάν. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ για να μας κάνετε αυτή την παρουσίαση και τώρα θα περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, την όθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε, ε, σε σχέση με τα έκθεση πρωτοβουλίες του κύριου Χέτμαν. Και στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης έδωσε έμφαση ο συγκητής στις παραμεθέριες ε, περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, καλύπτουν το 13% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά έχουν μικρούς να παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης. Κύριε, συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Χέτμαν, ε, αλλά λόγω κάποιου θανάτου στην οικογένειά του δυστυχώς δεν μπορέσε να παρευρεθεί εδώ. Παρέμεινε στην Πολωνία και γι' αυτό δεν μπορεί να παρουσιάσει την έκθεσή του. Πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλία στο θέμα και στο κείμενο αυτό του κυρίου Χέτμαν γίνεται αναφορά στη συζήτηση αυτή. Ο κύριος Χέτμαν ε, προσπάθησε να συμπεριλάβει όσο δυνατόν περισσότερα στοιχεία από αυτή τη συζήτηση. Αλλά ιδιαίτερα σε εκείνο το τμήμα της έκθεσης είπε, εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να ε, εκπονηθεί μια ξεχωριστή έκθεση για αυτές τις ε, εξόχως απόκεντρες ε, περιφέρειες. Ε, τώρα, στην έκθεσή του αυτή ασχολείται με τις 40 περιφέρειες εντό της Ελλάδας, ε, της, συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά είπε ότι πρόκειται να προτίθεται να συμπεριλάβει τις συμπληρωματικές τροπολογίες στην έκθεσή του. Η Επιτροπή στις 23 του 2017 εξάδωσε μία ανακοίνωση με το θέμα αυτό και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια τα οποία παρακολύουν την ανάπτυξη των περιφερειών αυτών. Η Επιτροπή έχει την άποψη ότι μπορούν να, αρθούν, να αρθεί ένα 20% των εμποδίων αυτών. Και με τον τρόπο αυτό το... θα, θα υπήρχε μία... Η έκθεση χωρίζεται σε τρία τμήματα. Στο πρώτο τμήμα ε, προσπαθεί ο εισηγητής μίσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα το επιχειρηματικό περιβάλλον να διαμορφώνεται αρνητικά. Ε, υπάρχουν διάφορα τέτοιου είδους εμπόδια, όπως υπόθηκε ήδη, και μεταξύ των εργαζομένων συχνά υπάρχει το πρόβλημα ε, της αναγνώρισης των πτυχίων και των διπλωμάτων, πώς θα ρυθμιστεί αυτή η αναγνώριση. Επίσης, κοινωνική ασφάλιση, το φορολογικό σύστημα κλπ. Ε, ε, μπορούν να οδηγήσουν σε διάφορα εμπόδια. Άρα η νομοθεσία όσον αφορά τις δημόσιες ε, δαπάνες, την κοινωνική ασφάλιση κλπ. θα πρέπει να ενοποιηθεί, να ομογενοποιηθεί. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια σχετική ρύθμιση, ούτως ώστε να βρεθεί ένας ή δυνατόν ένας κοινός παρανομαστής θα πρέπει να υπάρχει ε, μεγαλύτερη ευελιξία, αύξηση της εμπιστοσύνης και επίσης να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα γιατί η σημασία της ε, εκπαίδευσης και της πολυγνωσίας ε, στις παραμεθόριες αυτές περιφέρειες τονίζεται ιδιαίτερο στην έκθεση αυτή. Επίσης ζητήματα μετανάστευσης, τόσο στον τομέα της απασχόλησης, καθώς και στον το ζήτημα των ε, προσφύγων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μέρημνα ούτε ώστε το τοπικό επίπεδο να μπορεί να συνεργάζεται με το περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Στο τομέα της υγείας θα πρέπει να γίνει η προσπάθεια να υπάρξουν παροχές ε, διασυνοριακά. Ο τρίτος τομέας είναι η μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προγράμματα ραρκής συνεργασίας ε, ή ε, αυτό το οποίο προτίθεται να κάνει η Επιτροπή, δηλαδή να ε, συνεχίσει τα προγράμματα αυτά μετά το 2020, ούτως ώστε να μπορέσουν να αρθούν οι γραφειοκρατικοί φραγμοί και να μπορέσουν να αξιοποιηθούν τα προγράμματα αυτά. Γιατί μέσως λέγεται ότι οι πόροι οι οποίοι διατίθενται τελικά δεν απορροφώνται και όπως ε, υπόθεση τροπολογιών. Και εγώ από τη δική μου πλευρά θα ήθελα να πω ε, τρεις ε, φράσεις. Και εγώ λόγω των πρακτικών παραδειγμάτων, γιατί προέρχομαι από τη Σλοβενία, από μια περιοχή κοντά στη σύνορα με την Αυστρία και πολλά που αναφέρονται στην έκθεση. Παλαιότερα στην Αυστρία ε, θεωρούσαν ενοχλητικό για παράδειγμα να μιλάει κάποια σλοβενικά ενώ σήμερα δουν ε, οι προστατευτικοί ε, φραγμοί στην, στις κοινωνίε κοινωνίες ή όσον αφορά την κοινωνική προστασία για παράδειγμα μας κατέδειξε και πάλι και μιλώ για την οδό των Βαλκανίων από την Ελλάδα μέσω Μακεδονίας, Κροατίας, Σλοβενίας, αυτή σωστή συνεργασία και στις παραμεθόριες περιοχές. Σας ευχαριστούμε. Ήταν πολύ δύσκολο να διαβάσει κανείς ε, παρά τα πράγματα γιατί έχω iPad οπότε η οθόνη φωτίζεται από μόνη της. Δεν έχω άγραφο. Ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή για την παρουσίαση του σχεδίου έκθεση, γιατί πραγματικά δύσκολο πολλές φορέ οι συνοριακούς εργαζομένους να έχουν πρόσβαση σε καλύτερε μεταφορέ μεταφορές ή καλή υγειονομική περίθαλψη. Θα πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν τις υπηρεσίες όπως την αστυνομία και την πυροσβεστική που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των πολιτών. Επίσης, να τονίσουμε ότι τα Επίσης θα πρέπει να δώσουμε κάποια οικονομικά κίνητρα στις περιφέρειες που έχουν ε, σημαντικά βήματα διασυνοριακής συνεργασίας και ε, θα πρέπει να ε, στελεχώσουμε τις θέσεις εργασίας. Επίσης θα πρέπει να φέρουμε σε επαφή τις διασυνοριακές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της... Ε, οπότε, εκτός από τις εσωτερικές παραμεθόριες περιφέρειες, θα πρέπει να εκπονήσουμε μια στρατηγία της θαλάσσιας παραμεθόριες, εξωτερικές παραμεθόριες περιοχές της Ένωσης. Και θα πρέπει να ενταχθούν ε, ενεργά στην ε, διαδικασία ολοκλήρωση Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ με την σχετική πρόταση του Μίλη. Θα πρέπει να στηρίξουμε περισσότερο τα κράτη-μέλη στις προσπάθειές τους γιατί θα έχουμε επιθυμητά αποτελέσματα μόνο με συντονισμένο έργο σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό. Και θα πρέπει να καταρτήσουμε ένα συγκεκριμένο κατάλογο προτεραιοτήτων που αντιπροσωπεύουν 2% του καθάριστου ΕΠ, 200 21 ε, δισεκατομμύρια ευρώ και επίσης ε, θα διευκολύνουμε με τέτοια μέτρα την καθημερινότητα 150 εκατομμυρίων πολιτών που διαβιούν σε τέτοιες παραμεθόριες περιφέρειες. Γι' αυτό προσβλέπω σε αγαστή συνεργασία στο μέλλον. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστούμε κύριε Πίτσουλα. Από τις άλλες τώρα πολιτικές ομάδες δεν βλέπω κάποιο σκιώδη εισηγητή. Um, Οπότε να περάσουμε στο δεύτερο γύρο της συζήτησης με, το, όλα τα μέλη της Επιτροπής, και δεν έχουμε άλλους. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεση που εκπώνησε για τις παραμεθόριες περιφέρειες και εγώ ζω σε μια τέτοια περιοχή, 5-10 χιλιόμετρα, από δύο-τρία σύνορα χωρών και δική μου περιοχή εξοπεί ιδιαίτερως τα χρήματα, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής ε, όταν συζητούμε κατά πόσο είναι ουσιαστικά τα προγράμματα αυτά, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπει χρήματα για την ε, συνέχιση αυτών των προγραμμάτων και αυτό πραγματικά μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Ε, 9,5 δισεκατομμύρια για το διάστημα από 20 25. Πρόκειται λοιπόν για μια σημαντική αύξηση γιατί για το προηγούμενο διάστημα ήταν 6,6 δις. Άρα λοιπόν είναι πολύ καλό ότι αναγνώρισε η Κομισιόν αυτή την προτεραιότητα και αυτό είναι συμπολογισμό. Ε, και υπάρχει ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει εταίρως στους ανθρώπους πολίτες της παραμαθόριας περιφέρειας, και κάθαρο ποια χώρα είναι αρμόδια για θέματα υγείας στις παραμεθόριες περιοχές και ποια χώρα είναι αυτή η οποία καλύπτει τα έξοδα. Ε, υπάρχει το εργαλείο ΖΟΑΣΤΕ πλέον σουν ε, τα σύνορα, να προστρέξουν σε υπηρεσίες άλλες χώρες και είναι οι χώρες μεταξύ τους αυτές οι οποίες ρυθμίζουν το θέμα. Ε, και αυτό το ΖΟΑΣ περιγράφεται πολύ καλά στην Επιτροπή ως ε, best practice, βέλτιστη πρακτική. Οι ίδια να υιοθετήσουν το ΖΟΑΣ ε, γιατί είναι πραγματική ευλογία για τους Ευρωπαίους πολίτες των παραμεθόριων ε, περιφερειών. Και ένα δεύτερο εργαλείο που προτείνει η Επιτροπή είναι οι Ευρωπαϊκές Συνοριακές Συμβάσεις ε, δηλαδή εκ μέρους της επιχώρας να είναι εφαρμοστέο ε, στα, στα, στα, διάφορα προγράμματα. Ε, και με τον τρόπο αυτό θα διευκολυθούν πολλά προγράμματα και πολλές διασυνοριακές δραστηριότητε. Και θα ήθελα να παρακαλέσω την Επιτροπή ω τροπολογή στην λόγο έκθεση του κυρίου Χέτμαν ούτως ώστε να γίνουν τα πράγματα πιο συγκεκριμένα. Και αν δεν θέλει κανείς να πάρει το λόγο άλλο συνάδελφος, θα δώσει το λόγο στον κύριο Μπόγκοβιτ ή στην Επιτροπή μάλλον, ούτε ώστε να τοποθετηθεί εφόσον το επιθυμεί. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χωρίς φως και χωρίς φωνή δεν θα τα πάμε και πολύ καλά. Είμαι η Νάταλη Βόρσκελ από τη Γενική